και όχι να συγκροτήσουμε νέε, αλλά προτιθέμεθα να συζητήσουμε σε βάθο ε, την μελλοντική οργάνωση των εργασιών μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επίτροπε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ντερόσα, τον εισηγητή μα. Συνάδελφοι, έχω και καλά νέα. Ε, φτάσαμε στην τελευταία έκθεση για σήμερα. Ε, η έκθεση του κυρίου Κάτσμαντρικ, αντίκτυπο τη αναπτυξιακή πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η έκθεση που θα ψηφίσουμε αύριο είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης διότι τον Οκτώβριο η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα ανακοινοθέν για τις μελλοντικές προτεραιότητες των πολιτικών της. Επίσης θα παρουσιάσει και ένα σχέδιο για την συνεργασία. Στη Νότιο Κορέα θα έχουμε ένα φόρουμ υψηλού επίπεδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και αυτό το φόρουμ θα αποτελέσει και προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μπορέσει και το Κοινοβούλιο να παρουσιάσει τις δικές του προσδοκίες για την πράσινη βίβλο, την ανάπτυξη, την ενταξιακή και η φόρο ανάπτυξη. Εμείς όπως και ο Επίτροπος Πίβαλ θεωρούμε ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να στοχεύει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρέπει να αποφύγουμε μία κατάσταση ε, όπου θα συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στις λεγόμενες εύκολες χώρες, δηλαδή τις χώρες εκείνες όπου πριν βλέπουμε γρήγορα αποτελέσματα. Εμείς πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις χώρες εκείνες οι οποίες είναι πιο προβληματικές, οι οποίες είναι δύσκολες χώρες και να βοηθήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι υπόκεινται την διακυβερνησία. η αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει να διακόπτεται όταν μια φτωχή χώρα ε, περνάει στην κατηγορία των αναπτυσσομένων χωρών διότι ε, η περισσότερη, το μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας βρίσκεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θέλουμε η κάθε χώρα που δικαιούχος να αξιοποιείται πλήρως. Πρέπει να συγκεντρώσουμε τη βοήθεια στη γεωργία και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτούς τους τομείς το δυναμικό των αναπτυσσομένων χωρών είναι το μεγαλύτερο. Θα πρέπει η βοήθεια να στοχεύει στους στοχότερους και θα πρέπει να δεσμεύσουμε στις προσπάθειές μας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουμε και τη δράση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δύο άλλα σημαντικά πράγματα είναι η αηφόρος ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή. Όμως η συζήτηση που έδωσε και την πιο επόδυνη συζήτηση στην Αρπησιακή Επιτροπή ήταν ο όρος της ενταξιακής ανάπτυξη. Μην φοβόμαστε αυτόν τον όρο, διότι είναι η ανάπτυξη που εξισώνει τις κοινωνικές ανισότητες, είναι υπέρ των φτωχοτέρων. Και αυτού του είδους η ανάπτυξη πρέπει να είναι προσβάσιμη για τους φτωχούς και όχι μόνο για τους, ε, για τους ε, πιο ε, ενεργούς θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην εργασία, να βελτιώσουμε τις προδιαγραφές, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλειας και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα. Η Επιτροπή Ανάπτυξης επανέλαβε πολλές φορές ότι όταν ορίζουμε νέους, νέα καθήκοντα δεν πρέπει εμείς να ξεχνάμε και τις παλιές μας υποχρεώσεις. Και αυτή τη φορά θα πρέπει να κρατήσουμε τις υποσχέσεις του παρελθόντος. Είναι ηθική μας ευθύνη αλλά και παίζεται και η μας. Η αποτελεσματικότητα στην αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόσχημα για να παγώσουμε τη βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δράση μας και ευχαριστώ και όλους όσους με βοήθησαν για να συντάξω την έκθεσή μου. Ευχαριστώ κύριε Κάτσμαρκ. Κανείς δεν θέλει το λόγο. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ ε, και τον εισηγητή. Το θέμα της αύξησης ε, του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής ε, είναι ε, πολύ σημαντικό και η διακήρυξη του Παρισιού νομίζω ότι ακολουθεί τη σωστή προσέγγιση για να είναι πιο αποτελεσματική η αναπτυξιακή μας βοήθεια. Δεν θα πρέπει όμως να κάνουμε τη σύγχυση μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας και απόδοσης για τα χρήματά μας. Ο αριθμός σχολείων που χτίζουμε δεν είναι ταυτόσιμος με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο εν λόγω σχολείο. Και δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του να ζητάμε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα τα οποία δεν θα υποστηρίζουν καν του μακροπρόθεσμου στόχου για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη χρειάζεται χρόνο. Λυπάμαι αν αυτό δεν ε, συμβαδίζει με, τα με τις εκλογικές φιλοδοξίες του καθενός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το πλαίσιο κρίσης μας οδηγεί να ξανασκεφτούμε όλοι μας την δουλειά, στην αναπτυξιακή πολιτική για να βελτιώσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια και την, με μεγαλύτερη αποτελέσματα και την καταπολέμηση της στόχιας. Χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο συντονισμό της κοινοτική ενίσχυσης και των κρατών μελών. Και έχουμε τώρα την ευκαιρία να διπλασιάσουμε την προσπάθεια για τη βοήθεια γιατί ξέρουμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια από μόνη της δεν επιτρέπει να ξεριζώσουμε τη φτώχεια. Θα χρειαστεί να δώσουμε απάντηση σε διεθνές επίπεδο, όπως επίσης και αναθεώρηση των προτεραιοτήτων μας στο μέλλον έχουν ως εξή. Για, για τα σχέδια της χιλιετίας, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για να, να τελειώνουμε με τη φτώχεια. Δεύτερο, πρέπει να βρούμε νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Εμείς ξέρουμε ότι χρειάζεται αναπτυξιακή βοήθεια επισήμω, αλλά δεν αυκεί μόνη της για να ξεριζώσει τη φτώχεια. Θα πρέπει να έχουμε, να έχουμε να εισάγουμε το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα πρέπει να έχουμε μία ολοκλήρωση του σχεδιασμού για κατά της φτώχειας παράλληλα με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Στις αναδυόμενες χώρες θα πρέπει να αναπτύξουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας δίνοντας όμως αναπτυξιακή βοήθεια στις φτωχότερες χώρες για να φτάσουν αυτά τα επίπεδα. Η κυρία Ροήτοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, είναι ένα από τα στοιχεία ε, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και χαίρομαι που ο συνάδελφος κ. Κάτσμαρεκ έχει ακολουθήσει μια ελεύθερη προσέγγιση, όχι άκαμπτη προσέγγιση. Πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος ε, των μέσων και καλύτερη διαφάνεια για να αποφεύγουμε την διαφθορά. Επίσης, ε, ε, καταλαβαίνω τους φόβους του και τις ανησυχίες του ότι μπορεί να ε, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στις χώρες που είναι περισσότερο ασφαλείς, αποφεύγοντας τις χώρες που αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι χώρες που, όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ενδέχεται να είναι οι χώρες που χρειάζονται περισσότερο την αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης, στο σημείο 84, θέλω να τονίσω την ε, βαθιά μας ανησυχία για την αγορά γεωργικών εκτάσεων από ξένους επενδυτές, όπως από Κινέζους επενδυτές και αυτό υπονομεύει την τοπική επιστηστική ασφάλεια και ενδέχεται να έχει απρόβλεπτες ε, συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Φερέιρα. ανάμεσα στους στόχους αναπτυξιακής πολιτικής και τις συγκεκριμένες δράσεις που εφαρμόζονται υπάρχει μεγάλη απόσταση. Αναγνωρίζω τη σημασία της γεωργίας, της βιομηχανίας, ε, της ε, μεταφοράς γνώσεων, ε, τεχνογνωσίας. Είναι βασική παράγοντες ούτως ώστε να χειραφετηθούν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Αφετέρου όμως προκρίνουν όλη την απελευθέρωση του παγκοσμίου εμπορίου και τεχνοτοπιστωτικού συστήματος. Όμως αυτό τι σημαίνει για τις χώρε δεν έχουν αναπτυξιακέ δυνατότητε και υποτάσσονται όλο ένα και περισσότερο. Αναγνωρίζω πόσο σημαντικέ είναι οι δημόσιε υπηρεσίε ε, τη παιδεία ε, και την καταπολέμηση τη φτώχεια, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δέχονται απίστευτη πίεση από τα ε, διαρθρωτικά προγράμματα που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε διάφορε χώρε και τελικά δεν υπερέχει το δημόσιο συμφέρον, αλλά επικρατεί ήδη διπλωματία και όπως ακριβώς στον καιρό της απεικιοκρατίας και είναι ένας απλός παραλογισμός. Σας ευχαριστούμε. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, modernizácia európskej rozvojovej politiky musí nevyhnutne vychádzať z hodnotenia doterajších spôsobov fungovania rozvojovej politiky Európskej únie. Ο κύριος Πάσκα, κύριε Πρόεδρε, κύριε είναι σημαντικό να τονίσουμε τον αντίκτυπο της αναπτυξιακής πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει ε, να υποστηρίξει τα ε, ήθη και τις εργασιακές συνήθειες στις χώρες τις οποίες υποστηρίζουμε, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν ε, στο νέο σύστημα ε, να περάσουν από την προηγούμενη κατάσταση σε μια κατάσταση απασχόλησης ε, σε τομείς που είναι χρήσιμοι για την κοινωνία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και η φορολογική νομοθεσία να είναι δίκαια και πρέπει να διδάξουμε στους ανθρώπους αυτούς πώς να ψαρέψουν αντί να τους δίνουμε ψάρια όπως είναι η γνωστή αρχή. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχουμε λίγο χρόνο ώστε να μην καταλήξουμε στα μεσάνυχτα. Οπότε έχετε εσείς την επιλογή αν θα μιλήσετε γρήγορα ή αργά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Κατσμαράκη. Είναι μια συζήτηση πολύ επίκαιρη στο πλαίσιο των σκέψεων για τη μελλοντική πολιτική και η συζήτηση αυτή εντάσσεται πάρα πολύ καλά στα όσα ολοκληρώσαμε για την Πράσινη Βίβλο για την πολιτική ανάπτυξη Έχουμε 240 γραπτές απαντήσεις ε, καθώς ε, και πολλές παρεμβάσεις από ε, πολλούς ενδιαφερομένους και μπορείτε στην ιστοσελίδα μας να βρείτε αυτά τα στοιχεία. Έχοντας σκεφτεί τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα συντάσσει ένα ψήφισμα στη συνέχιση όλων αυτών, το οποίο θα ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί στα μέσα Οκτωβρίου βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων σε σχέση με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο της αναπτυξιακής πολιτικής. Συμφωνούμε ότι είναι ζωτικός ο ρόλος της ανάπτυξης σε αυτή την προσπάθεια. Ε, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις προτάσεις ε, της Πράσινης Βίβλου για την ενέργεια και για την επιστηστική ασφάλεια. Επίσης, συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο, όπως αναφέρεται στην έκθεσή σας, για τη ζωτική σημασία που έχει η σωστή διακυβέρνηση για τη μείωση της φτώχειας και για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επίσης ε, τονίζουμε παράλληλα και τη σημασία της σωστής λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων. Επίσης, ε, ο ρόλος της αναπτυξιακής βοήθειας μπορεί να βοηθήσει την πολιτική μεταρρύθμιση και αυτός είναι ένας ρόλος τον οποίο παίζουν τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια. Επιπλέον, Θέλουμε να συνεχίζονται ε, οι ενέργειες στον τομέα ε, ε, της ανάπτυξης και της ανάπτυξης ανθρωπινών πόρων και θα πρέπει να μην έχουμε στενό προσδιορισμό του εισοδήματος, αλλά να έχουμε ένα ευρύτερο προσδιορισμό των μέσων για την καταπολέμηση της φτώχειας. Συμφωνούμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια και όλοι είμαστε ικανοποιημένοι διότι το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευση των κρατών μελών να αυξήσουν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,7 του ΑΕΠ και Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρότασή σας, ιδίω στο σημείο, νομίζω ότι είναι το 49, ε, στο οποίο ε, μιλάτε για την ε, μετανάστευση και για την σύνδεση της εξωτερικής με την εσωτερική διάσταση της πολιτικής για την μετανάστευση. δεν θα εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στις αποκαλούμενες εύκολες χώρες, αποφεύγοντας τις χώρες που αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο, γιατί εκεί μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξη. Θα λάβουμε υπόψη μα τις προτάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Ακόμη τα σημεία τα οποία αναφέρεται για την ισότητα των φύλων είναι σημεία τα οποία θα λάβουμε υπόψη μας. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο εισηγητής κ. Κασμαρέκ θα, θα βρουν πολλές ε, ιδέες της έκθεσής σας οι οποίες συμπεριλαμβάνονται και στη δική μας ανακοίνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και σας κύριε Πρόεδρε και όλους τους βουλευτές. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που είχατε την υπομονή να μείνετε μαζί μας μέχρι τέτοια ώρα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάσμαρεκ, για την έκθεσή σας. Τώρα λοιπόν ολοκληρώθηκε και η συζήτηση για την έκθεση Κάσμαρεκ και πριν κλείσουμε έχω κάποιες ανακοινώσεις, θα τα διαβάσω στα τσεχικά. Ο Βίκτορ Σπάσκης μου μίλησε για τις ε, τελευταίες εξελίξεις και μου έχει στείλει